E, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ε, σημερινή σύνοδο, κυρίσω την έναρξη. Θέλω να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Φων Ρόμποϊ, να καλωσορίσω επίσης τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Επίτροπο που είναι μαζί μας. Και να περάσουμε στο πρώτο σημείο τη μερική διάταξη για σήμερα, που είναι τα συμπεράσματα από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Φομ Ρόμπο. Κύριε Πρόεδρε. Mr. President, uh, President of the Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι βουλευτές. Μέσα σε 49 ημέρες προέδρευσα τριών συνεδριάσεων